no hay anuncios y pasamos vale. directamente. Y aquí tenemos la lista de, de oradores. Sí. De oradores. Sí. Muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a esta comisión. Carlos Carlos. Καλώς... Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ε, του Προέδρου και θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, τον οικονομικό διάλογο δηλαδή, με τον Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, τον κύριο Λουίς Ντεγκίντος. Θέλω να ζητήσω συγνώμη για την απουσία της Προέδρου που δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την διαθεσιμότητά του σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουν δείξει όλοι οι Υπουργοί του Eurogroup αυτή τη διαθεσιμότητα. Ε, τον ευχαριστούμε. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δείχνει την επιθυμία της κυβέρνησης ε, την οποία εκπροσωπεί ο Υπουργός να συνεργαστεί με την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταία έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά από την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών πριν λίγους μήνες Ε, υπήρχε θέμα πάντα για τις συζητήσεις, στις συζητήσεις με την Ισπανία. Αλλά χωρίς ε, καθυστέρηση θα δώσουμε 15 λεπτά στον Υπουργό για να πάρει το λόγο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας. Presidente. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου που για δεύτερη φορά παρευρίσκομαι στην Επιτροπή σα. Πριν από ένα χρόνο, λίγο παραπάνω, ήμουν εδώ πάλι και σας ενημέρωσα για την οικονομική πολιτική την οποία αναπτύσσαμε στην ε, Ισπανία. Θα θυμάστε ότι τότε είχαμε μιλήσει για ένα πολύπλοκο σενάριο που αντιμετώπιζε η Ευρωζώνη εν γέννη. Είχαμε μια γενική οικονομική επιβράδυνση, είχαμε κρίση εμπιστοσύνη. Σήμερα η κατάσταση όπως είπε και ο Πρόεδρος, πριν διαφέρει σημαντικά. Πολλές από τις προκλήσεις τις έχουμε υπερβεί και μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα στο δεξιό το μέλλον. Η Ευρώπη δεν είναι πλέον η αιστεία και το επίκεντρο ανησυχιών που μεταδίδονται και σε αναδυόμενες χώρες. Πλέον η συζήτηση επικεντρώνεται σε ό,τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να έχει ποσοστά ανάπτυξης και να έχει και οικονομική ανάκαμψη. Είναι μεγάλη η πρόκληση αυτή για τους Ευρωπαίους ε, και την αντιμετωπίσαμε την κρίση με αποφασιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν και πρωταγωνιστή σε αυτή την ανάκαμψη και στη σημαντική προσπάθεια αλληλεγγύης και ολοκλήρωση που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προσπάθεια η Τραπεζική Ένωση είναι το σημαντικότερο βήμα που έχει κάνει η Ευρώπη μετά την εισαγωγή του ευρώ και θα αποτελέσει και ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία θα βασιστεί η ανάκαμψη ε, στην Ευρωζώνη. Εγώ πιστεύω ότι Ξεπεράσαμε τεράστια εμπόδια. Το 2014 επιτέλους είναι το έτος της ανάκαμψης. Το Νοσματικό Ταμείο επιτάνω έχει αναθεωρήσει τις προπικές ανάπτυξης της Ένωσης. Το 1% ωστόσο παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φτάσουμε στα επίπεδα ευημερία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την κρίση. Η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό τη, την ορμή τη και να συνεχίσει να εργάζεται για να γίνει μια πιο ευημερούσα, ισχυρή, ενωμένη Ευρώπη, αλλά με τι ίδιε ε, τι παντοτινέ τη αξίε. Με αυτή την έννοια είμαι βέβαιο ότι αυτοί οι οικονομικοί διάλογοι αποτελούν πάρα πολύ ε, σοβαρό στοιχείο αυτού του ε, ευρωπαϊκού εξαμήνου για να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση κυβέρνηση την Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ισπανική περίπτωση συγκεκριμένα. Πριν από ένα χρόνο ήταν πολύ διαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμασταν. Η ισπανική οικονομία αντιμετώπιζε δεύτερη ύφεση μετά από την έναρξη τη κρίση. Κράτησε πέντε χρόνια αυτή η κρίση και σε κανένα οικονομικό έτος δεν είχαμε σαφή ανάκαμψη σε ε, ε, αναντιστοιχεία με τις άλλες βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες. Ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, καταστρέφονταν θέσεις εργασίας, ε, είχαμε ασφάλιστρα κινδύνου γύρω στα 450 βασικές μονάδες και σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα η Ισπανία είχε μόλις απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας Οικονομική Βοήθεια. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αφήσαμε πίσω μας την ύφεση και η ισπανική οικονομία αντιμετωπίζει το 2014 ε, με τελείως διαφορετικές συνθήκες και όρους από τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα έχουμε συνεχή οικονομική ανάκαμψη, ανάπτυξη, η οποία ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2013 και θα ενταθεί και φέτος. Το ΔΝΤ βελτίωσε τις προβλέψεις του για την Ισπανία για το 2014 και μάλιστα είμαστε η δεύτερη πιο ε, θετική πρόβλεψη στην ε, Ευρωζώνη. Έχουμε μια πρόβλεψη για αύξηση της άξιας του 0,7%. Προσεκτική είναι αυτή η πρόβλεψη βέβαια, αλλά ένα θεμέλιο αυτής της ανάκαμψης ήταν η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως γνωρίζετε όλοι σας, η Ισπανία ε, το πρόγραμμα, μάλλον ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας. Το ολοκλήρωσαμε επιτυχία, διότι επικεντρώθηκαμε στις δύο βασικές αιτίες που δημιούργησαν και τις βασικές ανισορροπίες, τις σωρευτικές αυτές ε, στην ε, ισπανική οικονομία στα καλά χρόνια. Το πρώτο ήταν υπερβολική ιδιωτικό χρέος του ιδιωτικού τομέα και το δεύτερο ήταν η χαλαρή χρηματοοικονομική εποπτεία και βλέπαμε και στον ε, χρηματοοικονομικό τομέα υπερβολές. Είχαμε δηλαδή μη βιώσιμα ποσοστά προς, ε, ανάπτυξης πάνω από το 20% κατά μέσο όρο και οδήγησαν αυτά βέβαια στη φούσκα των ακινήτων. Μία φούσκα η οποία δημιουργούσε κάποια έσοδα φορολογικά συγκυριακά που έκρυβαν ουσιαστικά την τρύπα των δημόσιων οικονομικών και έθεταν σκηνή την βιωσιμότητά τους. Ενώ ταυτόχρονα είχαμε πληθωριστικές ε, τάσεις οι οποίες οδήγησαν σε σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Όλες αυτές οι υπερβολές ε, φάνηκαν ξεκάθαρα όταν ε, ξεράγει αυτή η φούσκα των ακινήτων. Το χρηματοπιστωτικό πρόγραμμα τι επιτυχή ε, μέτρα έλαβε. Πρώτα απ' όλα ε, εισήγαγε διαφάνεια στην πραγματική κατάσταση των ισολογισμών και έπειτα ενισχύθηκε η εποπτεία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η εταιρική διακυβέρνηση των Ισπανικών ε, τραπεζών. Με το πρόγραμμα αυτό καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση του κλάδου σε χρόνο ρεκόρ και σε βάθο. Και πιστεύω ότι πλέον έχουμε να μιλάμε για ένα πριν και για ένα μετά στο χρηματοπιστωτικό μέτρη τη Ισπανία. Είχαμε αναδιάρθρωση, ανακεφαλαιοποίηση, εξυγίανση των τραπεζικών και και χρηματοπιστωτικών εργασμών εν γέννη, τα ταμιευτήρια έγιναν τράπεζε με επαγγελματικά πλέον όργανα διαχείριση πιο ανεξάρτητα από την πολιτική εξουσία και συνεχίζονται οι, τα σχέδια αναδιάρθρωση και η Ισπανική Αρχή Εξυγίανση ε, έχει ασχοληθεί σε δύο περιπτώσει με το θέμα αυτό. Βέβαια σημαντικό είναι να έχουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη δυνατότητά τους να εκδίδουν στις διεθνείς αγορές, όπως είναι η Μπάνκια, η οποία πρόσφατα προχώρησε στην έκδοση ομολόγων της τάξης του ενός ε, δις. Είμαι πεπισμένος ότι οι Ισπανικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ε, τις δοκιμές αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με επιτυχία. Μια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση για να αλλάξουμε νοοτροπία και για να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία μας ήταν η μεταρρύθμιση ε, της αγοράς εργασίας που εγκρίναμε το Μάρτιο του 2012. Ήταν ε, πάρα πολύ άκαμπτη και υπήρχε και ένα διτό σύστρας από την αγορά εργασίας και μπορεί να μην έπεσε το ΑΕΠ στη διάρκεια της κρίσης. Καταστρέψαμε όμως πάρα πολλές θέσεις, το 50% σε σχετικούς όρους από ό,τι η υπόλοιπη η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασία ξεκινά του καρπού. Το 2014 σταθεροποιήθηκε η αγορά εργασία. Για πρώτη φορά από τότε υπάρξε η κρίση. Πέρυσι είχαμε μικρότερο αριθμό ανέργων από το 2012. Επίση είχαμε μια άλλη θετική εξέλιξη το τελευταίο τρίμηνο του έτου και για πρώτη φορά μετά το 2008 αυξά, αυξήθηκε. Ε, αυξήθηκαν οι θέσεις ε, εργασίας και έτσι Έχουμε γενικά 1% ε, δημιουργία, μάλλον κατόφλη ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν αρκούν όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό λοιπόν εφαρμόζουμε και άλλες καινούργιες μεταρρυθμίσεις. Το Δεκέμβριο εγκρίναμε μέτρα για την ε, ελαστικοποίηση της μερικής απασχόλησης, γιατί είμαστε πίσω στον τομέα αυτό σε ό,τι Ό,τι αφορά την εργασιακή χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση. Εκεί συνοδεύτηκαν και με διαρθρωτικά μέτρα για απελευθέρωση των αγορών, των υπηρεσιών και των αγαθών. Ο εξορθολογισμός δημοσίου τομέα. Δώσαμε νέα όθηση στην πίστη. Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Έτσι θα επικαιροποιήσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας και το σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα παρουσιάσουμε τον Απρίλιο. Αυτή είναι οι βασική άξονες. Θα συνεχίσουμε επίσης ε, να βαθύνουμε στη μεσομική ε, πειθαρχία. Το φορολογικό σύστημα θέλουμε να το κάνουμε επίσης πιο απλό για να έχουμε ενότητα αγοράς και φορολογική ουδετερότητα. Να δημιουργήσουμε επίσης κίνητρα για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, Θα αναθεωρήσουμε το αυτόνομο σύστημα χρηματοδότηση, Θα προωθήσουμε αλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και θα συνεχίσουμε τη μετάδοση τη ενεργειακή αγορά και τη αγορά των μεταφορών. Τις επόμενε εβδομάδε θα εγκρίνουμε το νόμο για τις επαγγελματικέ υπηρεσίες, ε, προτρέχοντας, τα έλεγα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να ληφθούν κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά τα ε, ρυθμισμένα επαγγέλματα, εμείς, τα κλειστά επαγγέλματα. Εμείς πιστεύω ότι αποδεικνύουμε ότι αποδίδει μια πολιτική ισορροπημένη διαθετικές ε, μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση και έτσι καταφέρουμε να με τις ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες που είχαμε. Μειώθηκε το ε, δημόσιο έλλειμμα με προσπάθειες όλης της κοινωνίας και ξανά αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στην ισπανική οικονομία. Επίσης είχαμε κάποια μισθολογική μετριοπάθεια, ένα είδος εσωτερικής υποτίμησης με αποτέλεσμα να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα και να μειώσουμε και το μισθολογικό κόστος. Επίσης, ε, με, μειώσαμε τις τιμές ε, με αποτέλεσμα να ευνοηθεί η όλη διαδικασία, αυξά, αυξήθηκε το εισόδημα πίσω των ε, οικογενειών, ευνοήθηκε η ιδιωτική κατανάλωση. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας επίση βελτιώθηκε και ως ό,τι αφορά την υπερχρέωση των οικογενειών και των ε, επιχειρήσεων της Ισπανίας μειώθηκαν πάνω από 200 δις, φτάνουμε πλέον στο 200 περίπου του ΑΕΠ και αυτή είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί. Πέμπτον, είχαμε ε, και προσαρμογή των ε, τιμών των κατοικιών. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις ε, αδυναμίες της Ισπανική οικονομία, Θα φτάσουμε σε ικανότητα χρηματοδότηση γύρω στο 2%, οπότε θα είμαστε σε μια θέση καθαρού πιστωτή και έτσι θα μειώσουμε και το χρέος μας. Ε, το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ελπίση ε, θεωρεί ότι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πλεονάσματος ε, στο ζύγιο τρεχόμενο λογαριασμό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπτυξη για το 2014, εξωτερικός τομέας θα είναι ο βασικό μοχλός, πρόβλεψη ανάπτυξη για την εξαγωγή αγαθών για το τρέχον έτος σημαντικές, γύρω στο 6% θα είναι γέννη το ποσοστό. Επίσης σιγά σιγά θα έχουμε και καλύτερη εσωτερική ζήτηση με βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και περισσότερες επενδύσεις ε, στα καταναλωτικά αγαθά. Οι εισαγωγές ε, επίσης και φαλοχικών αγαθών αυξάνονται με ε, ποσοστά της τάξης του 20% τα τελευταία τρίμηνα. Τώρα, συνεπεί όλων αυτών των προσπαθειών η ισπανική οικονομία πλέον γίνεται αντιληπτή τελείω διαφορετικά. Έτσι βλέπουμε από καθίσταται η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών και στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην πραγματική οικονομία. Η Άμεσε ξένε επενδύσει ε, έχουν διπλασιαστεί ε, μέχρι τον Οκτώβριο. Πάνω από τα 23 δι ε, τα ξεπέρασαν. Είχαμε επίσημα σημαντικέ μειώσει του μέσου κόστους, έκδοσης, μετά την εισαγωγή του ευρώ και μέσα σε ένα μήνα στο πάνω το 16% των αναγκών του σε χρηματοδότηση, το δημόσιο τα κάλυψε. Και θα έχουμε και μία πολύ σημαντική εξέλιξη με ζήτηση πάνω από τα 40 δις. Τώρα, για να έχουμε πραγματική ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθεί η διαρθρωτική κατάσταση, να έχουμε διαρθρωτικές βελτιώσεις, να έχουμε εμπορικό εξωτερικό πλεόνασμα. Δεν είμαστε πια εστία ανησυχίας για την αμαξορρόπηση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Και ολοκληρώνοντας θα πω ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει προσαρμόσει και μειώσει τις βασικές ε, ανισορροπίες. Κάτι αν προηγουμένω στην πρόσφατη οικονομική μας ιστορία καταφέραμε ε, να ακολουθήσουμε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Ως ισπανική οικονομία φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές γιατί είναι ακόμα εύθραυστη η ανάκαυση και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ε, γυρίσουμε σε επίπεδα απασχόλησης και εισοδήματος πριν την κρίση. Θέλουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ροή πίστοση δανείων προ του δυναμικού τομεί οικονομίας και σε εξηγία, ε, σε που θα έχουν, μάλλον θα Πρέπει να λάβουμε μέτρα για να πάψει ο κατακρεματισμό των αγορών που επιμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαια πιο δύσκολη ανάκαμψη σε όσε χώρε έχουν πληγεί από την κρίση και οι χώρε αυτέ βέβαια έχουν κάνει και τη μεγαλύτερη ε, προσαρμογή. Γι' αυτό θεωρούμε ότι με την Τραπεζική Ένωση θα σπάσει αυτό ο βάλο κύκλο του κατακρεματισμού των αγορών και γι' αυτό θα αγωνιστούμε για να, τον, ε, για να προωθήσουμε την Τραπεζική Ένωση και η κοινωνία της Ισπανίας και η γενικότερα Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε τα μάλα στην ανάκαμψη γιατί με την κρίση αυτή ε, πλέον βελτιώθηκε η έννοια της αλληλεγγύης. Οι ε, Ευρωπαίοι κατάφεραν εκ νέου να βρουν το δρόμο και θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη συζήτηση. Σας υπενθυμίζω ότι κάθε βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερώτηση. Πέντε λεπτά. Θα ξεκινήσω με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Φεγιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς Να καλωσορίσω τον Υπουργό. Και να πω ότι σε αυτή την πενταετή θητεία που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούω επιτέλου καλές ειδήσει με χαρά. Απευθύνω λοιπόν θερμούς σιβηρικούς χαιρετισμούς στο πρόσωπό σας και μια ερώτηση έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε από την κρίση. Κρίση η οποία ξεπερνιέται με δυσκολίες. Για να μην επαναληφθεί λοιπόν αυτό στο μέλλον, θα πρέπει να αποφύγουμε και κάποια σφάλματα που διπράχτησαν. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η ανάλυση σας για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο στην Ισπανία. Ποια είναι τα σφάλματα που διαπράχθησαν και τι πρέπει να κάνουμε για να τα αποφύγουμε. Ε, δεύτερον, τραπεζική ένωση. Υπάρχει πρόταση του Συμβουλίου, διακυβερνητική μάλλον, έναντι της οποίας το Κοινοβούλιο έχει διαφοροποιηθεί. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν βλέπετε πιθανότητες για συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Επίσης μιλήσατε για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Θα μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες, τι θα κάνετε στην Ισπανία, τι σκοπεύετε για τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, τι μέτρα θα λάβετε. Για τις δε άλλες χώρες, για να ολοκληρώσω, και πάλι με ιβυρική προσέγγιση, γιατί η Πορτογαλία ετοιμάζεται να βγει από το μνημόνιο με την Τρόικα θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η θέση σας ε, σε σχέση με την Πορτογαλία. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια και νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερος να συγχαρούμε τους Ισπανούς, τον Ισπανικό λαό, την Ισπανική κοινωνία και τους Ισπανικούς θεσμούς εν όλο. Συμφωνώ πάντως μαζί σας ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική από αυτό που είχαμε πριν από δύο χρόνια. Ξεκινώ με την τελευταία σας ερώτηση για την Πορτογαλία. Και πρέπει να πω ότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η πορτογαλική κυβέρνηση καταβάλει μια ολόψυχη προσπάθεια να αντιστρέψει την κατάσταση της οικονομίας της Πορτογαλίας. Έχει μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, έχει προβεί σε ξεκάθαρες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και στους προσεχείς μήνες είμαι βέβαιος η Πορτογαλία θα μπορέσει να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης οικονομίας. Και η Πορτογαλία θα αποτελέσει ακόμη ένα success story. Ήταν δύσκολο ο δρόμος. Αντιμετωπίσαμε πολλές αντικσιότητες και εσείς όπω και εμείς. Αλλά είναι πολύ σημαντική η ανάκαμψη της Πορτογαλίας για την Ισπανία και Τούμπαλιν. Όσο καλύτερα πάει η Πορτογαλία, τόσο καλύτερα θα πάει και η Ισπανία. Όσο καλύτερα πάει η Ισπανία, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρει και η Πορτογαλία. Σα ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία. Γιατί και αυτό θα αποτελέσει σημαντική χείρα βοηθεία για την Ισπανία και βέβαια την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, λάθη του παρελθόντο. Νομίζω ότι η ζωή μας διδάσκει πιο πολλά για τα λάθη, από τα λάθη μας παρά από τα δικαιώματά μας. Η ανάπτυξη, η υπερβολική ανάπτυξη του δανεισμού ήταν ένα από τα κύρια προβλήματα που οδήγησαν στην ε, φούσκα του ε, χώρου του τομέα των ακινήτων και όταν άρχισε αυτή να σκάει είδαμε δυσκολίες στην Πορτογαλία, προβλήματα και στον τραπεζικό κλάδο, σημαντική μείωση στα φορολογικά έσοδα και ε, στασιμότητα στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτή είναι η εικόνα που ακολούθησε τα καλά χρόνια, αφού ξεκίνησαν οι δυσκολίες λοιπόν. Και έτσι ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμος πιστεύω γιατί θα μας προσφέρει πιστεύω καλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και κυρίως των ταμιευτηρίων στην Ισπανία που τώρα έχουν μετατραπεί σε τράπεζες. Ιδιαίτερα δεν θα πρέπει να δώσουμε σημασία σε έναν επιμέρους δικτύο ο οποίος καταγράφει τις ανισορροπίες σε μια οικονομία, εθνική οικονομία, δηλαδή το, ε, τις ανισορροπίες στο εξωτερικό ισοζύγιο. Δεν μπορούμε να έχουμε 10% έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο ή περισσότερο. Επίσης ε, μιλήσατε για τραπεζική ένωση. Και για να ολοκληρώνω θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει πιστεύω σε μια πολύ λεπτή ισορροπία με την πρότασή μας. Χρειάζεται ο καθένας να κάνει τις υποχωρήσεις του. Αποτελεί ένα καλό σημείο κίνησης η πρόταση. Και ασφαλώς και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να μελετηθούν με προσοχή. Πάντως έχουμε μια συμφωνία στην οποία όλοι έχουν κάνει τις υποχωρήσεις τους. Για τις δημοσιονομικές εξελίξεις, πολύ σύντομα μπορώ να σας πω ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αποταμίευση, να δώσουμε κίνητρα για την απασχόληση, την ενσωμάτωση της αγοράς, του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας και βεβαίως οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες προβαίνουμε, για, το, για τη φορολογία εισοδήματο ε, και την εταιρική φορολογία θα είναι ο περιορισμός της ε, φορολογίας για τις εταιρείες και το κλείσιμο ορισμένων ε, κενών που είχαμε τόσο στην φορολογία επιχειρήσεων όσο και στην, επιχείρηση, στην φορολογία ιδιώτων. Ο κύριος Αντωνίν Σάντσε, εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δεγκίντο για την παρουσία του εδώ και για την παρέμβασή του και για την επιθυμία του να συνεχιστεί ο διάλογος στα πλαίσια της νομισματικής πολιτικής. Η σοσιαλιστική ομάδα πάντα θέλει να υπάρξουν σωστές επιλογές στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα και θεωρούμε ότι έχουμε αρχίσει να ξεπερνάμε μία ύφεση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, έχει τραυματίσει την Ευρώπη και αντιμετωπίζουμε μια κρίση θα έλεγα και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Η κατάσταση στην Ισπανία είναι οριακή και φαίνεται ότι οδεύει προς μια κάποια αποκατάσταση. Δεν έχει ξεπεραστεί βέβαια η κρίση, με τέτοια ποσοστά ανεργίας δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για, τη χρέωση, για το χρέη και των οικογενειών και των επιχειρήσεων και διότι οι πολίτες έχουν τα ελάχιστα για να επιβιώνουν και όχι να μπορέσουν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Ε, η καταπολέμηση της ανεργίας είναι ένας βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής και γι' αυτό θα ήθελα ακριβώς να θέσω κάποιες ερωτήσεις για το τι θεωρεί ότι πρέπει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να είναι κίνδυνος και να μην τηρήσει τις ανηλυμένες τις υποχρεώσεις. Οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα τεθούν σε λειτουργία από το 2014 και στα πλαίσια αυτού που είπατε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτή τη στιγμή έχει 10 πόντους διαφορά η Ισπανία με την υπόλοιπη, είναι στο 36,8 ενώ η Ευρωζώνη βρίσκεται στο 46,8. Η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης, η χαμηλή, ε, τα χαμηλά ποσοστά του πληθωρισμού ε, ίσως θα μας, δεν μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε ακριβώς αυτό το λεγόμενο κυκλικό έλλειμμα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να υπάρξει και σωστή ενημέρωση για τα δημοσιονομικά μέτρα και στα πλαίσια του επίπεδου του φόρου εισοδήματος και στα πλαίσια του ΦΠΑ. γιατί μόνο μια βίαιη μείωση των δημοσίων δαπανών θα οδηγήσει ίσως και θα πρέπει να συνοδευτεί και από μέτρα βία σε σχέση με την αύξηση των φόρων σε άλλους τομείς. Το θέμα είναι τώρα και να συζητήσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Εγώ στην παρούσα φάση δεν θα ήθελα να περάσω σε λεπτομέρειες να πω ότι και στον τομέα της αγοράς εργασίας ε, ε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες όμως να προσανατολίζονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, γιατί αυτό έχει οδηγήσει στη μείωση των θέσεων απασχόλησης και την χειροτέρευση των συνθήκων εργασίας. Ποιοι είναι οι προσανατολισμοί λοιπόν της εργασιακής σας πολιτικής, ποιες είναι οι πολιτικές, οι ενεργές και στον τομέα της μισθολογικής πολιτικής, γιατί ξέρουμε ότι ο ΙΜΠΕΞ έχει μειωθεί ουσιαστικά κατά ένα σημαντικό ποσοστό και δεν ξέρω αν με αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να βγούμε με συγκροτημένο τρόπο από την παρούσα κρίση. Να περιοριστείτε παρακαλώ στα 5 λεπτά. Θα είμαστε λίγο ευέλικτοι αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε. Πράγματι είναι γνωστή η πορεία της ισπανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητας, πράγματι οι μεταρρυθμίσεις οι δημοσιονομικές είχαν έτσι και αλλιώς θετικές επιπτώσεις της οικονομίας, όπου είναι σαφές ότι το σύστημά μας δεν λειτουργούσε με σωστό τρόπο. μια μεταρρύθμιση δημοσιονομική μπορεί να ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Για πρώτη φορά η Ισπανία τώρα πλέον στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου δημιουργεί καθαρή απασχόληση. Eso, eh, sin duda, algo Είναι ένα θετικό, πάρα πολύ θετικό στοιχείο στον τομέα της απασχόλησης. Θα είναι μια καλή χρονιά για την απασχόληση στην Ισπανία φέτος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Τρεμόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρεις ερωτήσεις σύντομες. Η πρώτη. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, η μη... de más del 10%. Al mismo tiempo crece ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αρχίσει να δημιουργεί και αυτός προβλήματα και να επηρεάζει αρνητικά την οικονομική κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργείται επίσης και από την έλλειψη ροών πιστωτικών από τις τράπεζες και από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις. μετά από πάρα πολλά χρόνια ανεξέλεγκτου δημοσίου χρέους προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε τώρα. Τι προετοιμάζει η κυβέρνησή σας, απλά μεταρρυθμίσεις ή μόνο μειώσεις στον τομέα των δημοσίων δαπανών. Και θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει με το δημοψήφισμα στην Σκοτία και πόσο αυτό θα επηρεάσει τα πράγματα στον τομέα της οικονομίας στην περίπτωση κατά την οποία η Σκωτία επιλέξει τον δρόμο της ε, ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να ισχύσει κάτι αντίστοιχο και στην περίπτωση ενός θετικού αποτελέσματος ε, σε δημοψήφισμα στην Καταλωνία. Έχουμε περάσει από μια διαδικασία εξυγίανσης λοιπόν της ε, ισπανικής ε, ε, οικονομίας. Σε κάποιους τομείς τα πράγματα έχουν πάει υπάρχουν πολλές νέες επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ενδείξεις για νέες πιστοτικές θετικές ε, ροές. Όλοι οι δείκτες τους οποίους έχουμε δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάκαμψη και στον τομέα της προσφοράς και στον τομέα της ζήτησης ε, σε επίπεδο ενυπόθηκων δανείων ή δανείων καταναλωτικών. Το θέμα είναι να υπάρχουν σωστά κίνητρα και στον τομέα των δημοσιονομικό έτσι ώστε να υπάρξουν κίνητρα και για τις επενδύσεις και για την αύξηση της απασχόλησης. Και σύμφωνα πάντα και με τους δείκτες και τις υποδείξεις και του ΟΣΑ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε σχέση με το τελευταίο θέμα το οποίο θέσατε, όπως γνωρίζετε στην παρούσα φάση, ε, τα οικονομικά πάρα πολλών ε, οικονομικών αυτόνομων περιοχών. Αυτό που δείχνουν είναι η μεγάλη δύναμη την οποία δείχνει συνολικά η χώρα, η Ισπανία. Όλοι μαζί ενωμένοι είμαστε πάρα πολύ ισχυροί και σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτή η ισχύ βοηθάει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και θέτει σε λειτουργία την αρχή της αλληλεγγύης και σε επίπεδο οικονομικών ε, επιτευγμάτων. Perdón, tengo un minuto de slot. Έχω ένα λεπτό ακόμη. Σα ευχαριστώ για τι απαντήσει σα. Δεν μου απαντήσατε όμω το τρίτο ερώτημα. πανική Ισπανική κυβέρνηση εγγυάται το δημόσιο χρέο σε περίπτωση δημοψηφίσματος. Ε, το 75% των Καταλανών ξέρετε στηρίζει το δημοψήφισμα ε, και τα κόμματα που είναι υπέρ του δημοψηφίσματος ε, κερδίζουν όλο και περισσότερε ψήφου. Ναι ή όχι λοιπόν. Απάντηση. Κοιτάξτε, η θέση τη Ισπανική κυβέρνηση σε σχέση με το δημοψήφισμα είναι απόλυτα γνωστή διαστόματος και του Προέδρου της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος κυβέρνηση τα έχει πει και σας παραπέμπω σε αυτά που έχει πει. Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα όμως που είπατε, η μόνη πηγή χρηματοδότησης για μια σειρά από αυτόνομε περιφέρειες μεταξύ αυτών και της Καταλωνία είναι το δημόσιο, το ισπανικό. Το Ταμείο ρευστότητα ε, και το Ταμείο Πληρωμών των Πιστωτών. Θα σας ε, παραπέμψω σε κάτι που είπα πριν, ότι δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει πλέον αλληλεγγύη μεταξύ των ε, αυτόνομων περιφερειών, καταδεικνύεται αυτό και με το Υπουργείο Οικονομικών. Για το Φεβρουάριο, για παράδειγμα, θα έχουμε τη δεύτερη πληρωμή προμηθευτών, τη δεύτερη προσπάθεια πληρωμής ε, των προμηθευτών από πλευρά Ισπανικής κυβέρνησης ε, και θα διατεθούν 8 ε, δις ευρώ το Φεβρουάριο στις αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας ώστε πολλές αυτόνομες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και που δεν είχαν πρόσβαση στην αγορά και δεν μπορούσαν να πληρώνουν τόσο ψηλά ε, επιτόκια και γιατί δεν είχαν κυρίως πρόσβαση στην αγορά βέβαια, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις βασικές θεμελιώδεις υπηρεσίες αυτό, το επαναλαμβάνω, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη και μεγάλη οικονομική ολοκλήρωση. Και το γνωρίζετε και εδώ στο Κοινοβούλιο και στα κοινοτικά θεσμικά όργανα, ότι γίνεται λόγο και αυτό το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανση των Τραπεζών και των ενιαίων οπτικών Μηχανισμό και τον ενιαίων Μηχανισμό Εξυγίανση. Αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό βήμα προ τα εμπρό αυτέ τι δύσκολε στιγμέ που αντιμετωπίζουμε. Και δει η οικονομική, ε, δημοσιονομική ολοκλήρωση και αυτή η αλληλεγγύη. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φίλιπ Λάμπερτ τώρα έχει το λόγο. Κύριε Δεκμήντος, καταρχάς ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σημειώνω την δεύτερη φορά που έρχεστε. Επίσης σημειώνω ότι ο ε, προσβοράν γειτονά σα, ε, Πιάχ έχει τρει ή τέσσερι φορέ απορρίψει πρότασή μα. Δεν ξέρω αν αυτό ε, οφείλεται στο ότι είναι πιο νεαρή δημοκρατία στην Ισπανία από ότι στη Γαλλία και είναι ίσω πιο ισχυρή ή πιο έντονο το αίσθημα τη λογοδοσία, Πάντω, σα ευχαριστούμε. Πιο σοβαρά πάντω, αν και η δημοκρατία είναι ήδη σοβαρό θέμα, με ανησυχούν ιδιαίτερω οι ανισότητε στην Ισπανία. Τι μπορείτε να πείτε λοιπόν σε όλου αυτού και ιδιαίτερα σε αυτούς που πληρώνουν το κόστο τη κρίσης στην Ισπανία. Αυτούς που προκάλεσαν την κρίση στην Ισπανία, διορθώνω. Αυτούς δηλαδή που ε, έσπρωξαν στην ε, φούσκα το, της αγοράς ακινήτων. Τραπεζίτες ε, και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πλήρωσαν τις συνέπειες της κρίσης γιατί αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν τελικά το λογαριασμό ήταν ε, εκείνοι που βρισκόνται στο κατώτερο οικονομικό επίπεδο. Η ανεργία είναι χειρότερη, οι ανισότητες, τα οικονομικά προβλήματα για όλους αυτούς είναι πολύ πιο σοβαρά. Έτσι λοιπόν, ναι, μπορεί να μπορεί σιγά σιγά να ε, επισκευάσει μέρος αυτής της ε, φούσκας η Ισπανία και μας λέτε ότι γίνεται πρόοδος σιγά σιγά, αλλά δεν βλέπω αυτοί που ωφελούνται από την ε, κρίση, μάλλον αυτοί που πληρώνουν την κρίση δεν είναι αυτοί που ωφελήθηκαν από την φούσκα. Τι θα μας πείτε λοιπόν, σε εμά και σε αυτούς. Απάντηση. Βεβαίως, ήδη στην παρέμβασή μου στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει επεσήμανα ότι υπάρχουν ανισότητε. Αυτό οδήγησε και στην κρίση και, στην, και η τραπεζική αστάθεια οδήγησε στην ε, φούσκα και με τη σειρά της αυτή σε όλα τα άλλα προβλήματα. Ο κύριος λόγος λοιπόν ύπαρξη αυτού του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ήταν ακριβώς να αποτρέψει τέτοιου είδους προβλήματα στο μέλλον. Στην η Ισπανία δεν κάναμε διάσωση τραπεζών. Κάναμε διάσωση, διάσωση ε, καταθετών. Και αυτό πρέπει να το θυμίζουμε πάντα γιατί καμιά φορά λησμονείται. Έχασαν οι μέτοχοι τα πάντα. Τροποποιήθηκαν ομάδες ε, διαχείρισης, ε, manager. Ορίσαμε αυστηρά ε, ανώτατα επίπεδα για τις αμοιβέ τους αυστηρά κριτήρια για την διακυβέρνηση των τραπεζών, διορθώσαμε τα προβλήματα που είχαμε σχέση με τα ταμιευτήρια και αποκαταστήσαμε πολλά άλλα προβλήματα στο τραπεζικό τομέα, στον οποίο οφείλονταν πολλά από τα προβλήματα. Αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να διοχετευθεί ε, κεφάλαιο στις τράπεζες, κάτι το οποίο ίσως είναι δύσκολο να εξηγηθεί πολλές φορές, αλλά είναι εναλλακτική θα ήταν πολύ πιο επώδυνη και δαπανηρή, γιατί θα οδηγούσε σε πολύ πιο σημαντική οικονομική κρίση και στην Ισπανία και βέβαια στασιμότητα ή πτώση στην οικονομική δραστηριότητα, πολύ σοβαρότερη από την πολύ ήδη σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Τούτου λεχθέντος, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε, όπως είπα και νωρίτερα, τα ασφάλματα του παρελθόντος, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και ανισορροπίες της οικονομίας της Ισπανίας, να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την εξέλιξη του ε, επίπεδου δανεισμού, του τρόπου δανεισμού, την εξέλιξη στις τιμές των ακινήτων, την ε, εξέλιξη στο εξωτερικό ισοζύγιο, στο εξωτερικό έλλειμμα και να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να ζούμε με χρέος χωρίς παραγωγικότητα, χωρίς αποτελεσματικότητα, χωρίς ανταγωνιστικότητα. Γιατί αυτές θα είναι οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομίας της Ισπανίας. Από την άλλη βλέπουμε κάποια πολύ θετικά βήματα στην ε, ισπανική οικονομία. Δεν ξέρω αν είδατε τι εικόνα παρουσιάζουν πλέον οι εξαγωγές μας, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μας ή η εξέλιξη των ξένων επενδύσεων, των επενδυτικών ροών προς την Ισπανία. Αυτό δείχνει ότι έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και προχωρούμε καλά. Εάν βέβαια με ρωτήσετε ποιο είναι το κύριο δίδαγμα που μπορώ να αντλήσω, το κύριο συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να καταλήξω από την κρίση αυτή και για τις τράπεζες, τα ταμιευτήρια και την αναδιάρθρωσή τους όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι η διαφάνεια και η σαφήνεια είναι ο κύριος μοχλός που θα κινήσει την οικονομία. Και πρέπει να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό εγχείρημα. Έχω πει ότι πέραν των κεφαλαιοχικών απαιτήσεων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής της, αυτού του εγχειρήματο. Ε, πέραν αυτών λοιπόν θα πρέπει να διασκεδάσουμε όποιες ανησυχίες και αμφιβολίες ως προς την υγεία των τραπεζών μας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο να εξασφαλίσουμε πραγματική ανάκαμψη εάν δεν είναι υγιές το τραπεζικό σύστημα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το ε, ισχυριστεί πλέον η Ισπανία ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα φερεγγιότητας του τραπεζικού της συστήματος. Και με τις εξελίξεις και στην Τραπεζική Ένωση πιστεύω πέραν της ε, προσπάθειας που έχει κάνει η Ισπανία ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τη σαφήνεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο κύριος Βίλι Μέγερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Έθατε εδώ για να πλασάρετε, να πουλήσετε το ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την οικονομική κατάσταση της Ισπανίας, αλλά δεν ανταποκρίνονται αυτά με την έκτακτη ε, κατάσταση που ζει η χώρα μας, που δεν την είχαμε γνωρίσει μετά τη δικτατορία σε αντίστοιχα επίπεδα. Εσείς στηρίζετε κάποιες πολιτικές που σε ουσιαστικά ε, σας τις δίνει η Τρόικα γραμμένες, ε, οι μισθοί, τα δημόσιες υπηρεσίες, οι συντάξεις πλήττονται. Και νομίζω ότι και στον ενεργό πληθυσμό βλέπουμε προβλήματα. Ε, υπάρχει μεν μείωση της ανεργίας, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο ότι έχει αυξηθεί η απασχόληση πάνω από 190.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν, αλλά χάνονται κάποια απλά από, τις, από τα στατιστικά στοιχεία. Ε, το 60,8% των σχεδόν 6 εκατομμυρίων ανέργων να ψάχνουν πάνω από ένα χρόνο δουλειά. Και εσείς έχετε ε, ακολουθήσει μια οικονομική πολιτική για να λύσετε με δημόσια κονδύλια τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η ιδιωτική διαχείριση του χρηματοπιστωτικού τομέα που σίγουρα ε, πρόκειται για μια οργανωμένη απάτη. Επιχειρήσεις, διαχείριση χρηματοπιστωτικού τομέα που είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας ε, να φτάσει σε ένα διέξοδο διότι οι εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, ε, οι πολίτες, γιατί να πληρώνουν το τίμημα για τις ε, απάτες που έκαναν όλοι αυτοί οι, οι και τα ξέρετε πολύ καλά από μένα. Γιατί για κάποιες επιχειρήσεις γνωρίζετε και εσείς ήσασταν, είχατε κάποια ε, συμμετοχή. Και όλη η αισιοδοξία σας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για πείτε το στους εργαζόμενους ε, από όλη την Ισπανική επικράτεια. Τα... Τις επιχειρήσεις που βάζουν λουκέτο, ε, τις οικογένειες, τα νοικοκυριά που δεν έχουν τίποτα, στηρίζονται στα προνοικά επιδόματα. Οι νέοι που φεύγουν και αυτή η πολυεθνική κοκακόλα που θα βγάλει στο δρόμο 742 στο στα Βαλιαρίδες, της Αστούριας, ε, σε άλλες περιοχές. Ε, ε, ποιο, τι σας κάνει να έχετε αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι 6 εκατομμύρια άνοιγοι περίπου δεν έχουν καμία συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν πρέπει να πληρώνουν ε, τους απαταιώνες οι πολίτες. Και ένα ερώτημα για να κλείσω. Μέρος του δημόσιου χρέους οφείλεται στην κερδοσκοπία. Η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να δίνει άμεσες ενισχύσεις, ε, αλλά δανείζει με επιτόκια στα συσοτικές τράπεζες που ε, τελικά με άλλα επιτόκια και τα λοιπά και καπέλα που βάζουν ε, καταλήγουμε σε κερδοσκοπία. Μήπως πρέπει να γίνει έλεγχος ε, ε λογιστικός για να δούμε γιατί μιλάμε, τι είναι αυτό το εξωτερικό χρέος. Εμείς έχουμε δεσμευτεί από πλευρά ΕΕ αριστερά στην Ισπανία και άλλα όμως ευρωπαϊκά κόμματα, γιατί θέλουμε να διευκρινίσουμε και να ξέρουν οι πολίτες μας γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για χρέο. Θέλω λοιπόν να υπάρχει ένα σαφή έλεγχο και να οριστεί τι οφείλουμε πραγματικά και τι είναι προϊόν κερδοσκοπία. Τέλο, ε, είσαστε και κάνετε, φέρετε σε πέρα στο ρόλο σας. Ουσιαστικά ε, επαναλαμβάνετε σαν ένα μάντρα, σαν ένα σύνθημα έτσι όλα αυτά, ε, ότι πηγαίνουν όλα καλά κτλ αλλά δέκα χρόνια φαίνεται ότι θα περιμένουμε για να έχουμε την ίδια δραστηριότητα ε, απασχόληση που είχαμε πριν από την κρίση. Και διαβάζω και τι δικέ σα ε, δηλώσει. Και ο Επίτροπο, ή ο άλλο Επίτροπο τέλο πάντων, ε, είπε ότι δεν αρκεί να βρει κανεί μια θέση εργασία για να μειωθούν οι ανισότητε. Δεν αρκεί έβριση μια θέση εργασία και θα ολοκληρώσω. Είναι νομίζω σαφής η πραγματικότητα και αφήστε, δεν υπάρχει καμία συγκρατημένη εξοδευτική απάντηση. Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος για συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε τρομερές δυνατότητες ε, στην ισπανική οικονομία. Σίγουρα υπήρξαν μεγάλες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Ε, μιλήσατε για ε, την απασχόληση και ότι πράγματι βγήκαν κάποιοι τον εργό πληθυσμό και δεν φαίνεται να είναι στην ανεργία. Ε, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε και με δυο μάτια τα πράγματα. Στο τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας στην Ισπανία. Πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό, όπως και εγώ αναγνωρίσω αυτά που λέτε. Α είμαστε αντικειμενικοί όσο μπορούμε. Τόσο ό,τι αφορά τον έλεγχο, οι Ισπανικέ τράπεζε εποπτεύονται από την Τράπεζα τη Ισπανία ε, ή θα εποπτεύονται σε λίγο καιρό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι σαφές τότε, θα είναι σαφές τότε ποια θα είναι η θέση τους ε, σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος. Τώρα, δεν ξέρω εσείς τι θέλετε. Να μην ε, υπάρχει χρηματοδότηση του δημόσιου ελλείμματος. Μήπως έτσι όμως θα φτάνουμε σε κατάρρευση των δημόσιων ε, υπηρεσιών στην Ισπανία. Δεν νομίζω να θέλετε κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι όμως μας τα παρουσιάσετε τα πράγματα. Μπορεί και να μην κατάλαβα τι θέλετε να μου πείτε βέβαια, να μην άκουσα καλά, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι λογικό ότι πράγματι βλέπουμε μια κατάσταση όπου οι ισπανικές τράπεζες έχουν ε, δημόσιο χρέος με τη βελτίωση ή τέλος πάντων συνεπία της βελτίωσης της όλης αντίληψης που είπα πριν όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει ότι μειώνεται το δημόσιο χρέο, μειώνεται το ποσοστό τέλο πάντων που είχαν στα διάθεσή του οι Ισπανικέ τράπεζε και η Ισπανική οικονομία πηγαίνει πολύ καλύτερα σε σχέση με ό,τι γινόταν πριν από δύο χρόνια. Και φυσικά και τα δημόσια ταμεία, το Υπουργείο Οικονομικών ε, πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε έκδοση ομολόγων. Ξέρετε τα ποσά, έχουμε και 23 δις για τη χρηματοδότηση των αυτόνομων περιφερειών και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι και η σπονδυλική στήλη του κράτους πρόνοιας. σε ευχαριστώ πολύ. όνομα του Ιευτή ο κύριος Στέρχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας για άλλη μια φορά. Χαίρομαι για τα συγκρατημένα καλά νέα που μας φέρατε και την ε, επιστροφή παραδείγματι στις αγορές της χώρας, αλλά υπάρχουν κάποια ε, προβλήματα ακόμη, παραδείγματι πολύ σοβαρά ε, χρέη στο ισοζύγιο των τραπεζών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πώς ε, μπορείτε να θεωρείτε ότι οι τράπεζες μπορούν να σταθούν στα πόδια τους μόνες τους χωρίς να χρειαστεί άλλη διάσωση. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι οι ισπανικές τράπεζες θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες και την ε, αναθεώρηση και το τεστ αντοχής που θα λάβει χώρα όπως προβλέπεται από την ε, ενιαία εποπτική αρχή. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο κύριος Χέκμαρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ισπανική οικονομία. Όλα αυτά είναι θετικά για την Ευρώπη. Είναι συνολικά καλό γιατί ανακάμπτει η ισπανική οικονομία αλλά και σε σχέση με την επιλογή των σωστών πολιτικών. Είναι άδικο λίγο και παράδοξο ότι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα είναι, ε, ε, υφίστανται περισσότερη κριτική από αυτούς που προκάλεσαν το πρόβλημα οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από τις συζητήσεις. Και ίσως να δημιουργείται και λανθασμένο μήνυμα σε σχέση με τις πιθανότητες των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε δύο επιλογές στο μέλλον. Είναι η, από τη μία υπάρχει αντίληψη ότι θα πρέπει να δαπανούμε όλο και περισσότερο και η μηχανή θα καλύπτει αυτές τις συνεχείς δαπάνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Πιθανώς εδώ να μην υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και από την άλλη η πολιτική είναι η, λιτότητα, αλλά δεν είναι σωστός όρος λιτότητα, είναι μεταρρύθμιση. Reformity λέει ο μιλητής. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε να εκτιμήσετε σε ποιο βαθμό τα προβλήματα της Ισπανίας χειροτέρευσαν από τις δαπάνες τις οποίες ε, είχε προβεί η κυβέρνηση Ζαπατέρο. Έχει μεγάλη αποφασίσει να λύσουν τα προβλήματα ξεπερνώντας τα προβλήματα και θυμάμαι και την αντιπολίτευση τότε το 2009 που έλεγε ότι και στη Σουηδία που έλεγε ότι ίσως θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε τα ίδια που κάνει η Ισπανία. Βέβαια το 10 δεν το έλεγαν πια αυτό. Γιατί είχε αποδειχθεί ότι η μέθοδος αυτή η Ισπανική δεν ήταν σε καμία περίπτωση η μέθοδος Ζαπατέρο σωστή. Πώς εσείς ε, λοιπόν επιδράτε την κατάσταση, ε, το τι είχε συμβεί τότε στην σημερινή κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να στραφώ στο μέλλον λέει ο κ. Δεγκίντος. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Η Ισπανία μπήκε ε, στην κρίση ήδη από το 2007. Τότε είχαμε ένα πλεόνασμα και ήμασταν 20 πόντους κάτω από τους, ε, από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αλλά τα φορολογικά κίνητρα τα οποία είχαμε δώσει και ε, στην Ισπανία ήταν τα πιο ισχυρά πόλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά όλα δημιούργησαν προβλήματα και το δημόσιο χρέος άρχισε να αυξάνεται. Το θέμα δεν ήταν μόνο η δημοσιονομική μας πολιτική μόνο. Το θέμα είναι ότι αγνοήσαμε εν πολλής ε, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί σε σχέση με ε, την σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό χρέος και τα πιστοτικά ιδρύματα. Στην ουσία εμείς κάναμε ότι δεν βλέπαμε ποια ήταν η πραγματική κατάσταση των τραπεζών και στην ουσία στο τέλος του 2011 η κατάσταση πλέον ξεπέρασε τα όρια και στις αρχές του 2012 και η κυβέρνηση έπρεπε σε τρεις μήνες να κάνει ό,τι δεν είχε γίνει σε τέσσερα χρόνια. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Η κατάσταση λοιπόν ήταν πάρα πολύ κρίσιμη. Καμία χώρα νομίζω δεν αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα όπως αυτά που αντιμετώπισε η Ισπανία. Όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα και μας διαφοροποιούν από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ε, δεν είχαμε μπορέσει να αναπτυχθούμε και να ανακάμψουμε το 2010 και το 2011. Ε, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπήρχε οικονομική ανάκαμψη εκείνη την εποχή και είχαμε και πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα της, ε, ε, των εργασιακών πολιτικών και της απασχόλησης. Η κατάσταση λοιπόν ακόμα και στην περίοδο 2007-2009 είδαμε ότι είχε αυξηθεί το δημόσιο χρέος μέσα σε μία πολύ μικρή περίοδο, μία διετή περίοδο. Το βασικό μάθημα λοιπόν το οποίο μπορεί κανείς να πάρει από εκείνη την περίοδο είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές και στις διαρθρωτικές αλλαγές και στις διαρθρωτικές ανισορροπίες που έχουν σωρευθεί. Απόλυα ανταγωνιστικότητας, υπερβολικό ιδιωτικό χρέος, ε, φούσκες στον τομέα των κατοικιών και της οικοδομής. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να διορθώσει τα προβλήματα μόνο μέσω δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον Υπουργό και να τον ευχαριστήσω για τις απαντήσεις και την παρουσίαση του. Ξεκινώντας θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ. Η κυβέρνησή σας μπόρεσε σε πολύ δύσκολες εποχές που ανέλαβε καθήκοντα να ξεκινήσει αμέσως τις μεταρρυθμίσεις των οποίων τα θετικά αποτελέσματα δύο χρόνια μόλις μετά την ε, ανάληψη των καθηκόντων της το δεύτερο τρίμηνο του 2013 άρχισαν να φαίνονται να γίνονται ορατά. Ξαναδώσατε λοιπόν εμπιστοσύνη στην οικονομία τη Ισπανία και βλέπουμε μια ανάκαμψη. Πολύ είναι οι λόγοι για του οποίου πρέπει να σα συγχαιρόμαστε. Αν και μένουν αρκετέ προκλήσει ακόμη, γιατί πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματο υγεία, να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ταξιδιωτικού η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασία. Όλα αυτά είναι μεγάλε προκλήσει που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνησή σα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω στον δρόμο αυτόν. Έχετε στήριξη και συνένεση στην Ισπανία. Και πώς εξασφαλίζετε εάν υπάρχει αυτή η συνένεση. Καλείτε επιχειρήσεις μη ε, κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών, τοπικές περιφερειακές αρχές για να εξηγήσετε και να εξασφαλίσετε συνένεση για τα μέτρα που σκοπεύετε να πάρετε και έχει βοηθήσει αυτό στην αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη τι μέτρα λαμβάνετε για τη δημοσιονομική εξυγίανση σε σχέση με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ποια μέτρα ήταν πιο βραχυπρόθεσμα και ποια ήταν τα πιο επώδυνα και σκληρά. Και σε αυτό θα δώσω έμφαση διότι αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και εμείς στην Κροατία με περικοπές εταίρως στις αμοιβέ και τις συντάξεις μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση φτώχεια, σε μείωση εισοδήματων και βέβαια αυτό δεν πρέπει να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για, τις, <laughs> για συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλη όκληρη την κοινωνία της Ισπανίας πρέπει να συγχαιρόμαστε. Η κυβέρνηση βέβαια είχε την ευθύνη της επιδίωξης των κατάλληλων πολιτικών, αλλά ολόκληρη η κοινωνία της Ισπανίας έχει συμβάλει σε αυτή την ε, επιτυχία και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και εμείς οι πολιτικοί, γιατί είναι δύσκολο μερικές φορές να εξηγούμε στην κοινωνία ότι κάποια μέτρα μπορεί να είναι πικρά, σκληρά, αλλά μπορεί να δώσουν τελικά ε, επούλωση στις πληγές της οικονομίας. Μπορεί να οδηγήσουν σε εξηγένσεις οικονομίας. Όμως ήταν, ε, νομίζω, όριμη η κοινωνία της Ισπανίας και επέδειξε ευφυΐα στο να αντιληφθεί ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να ξεφύγει από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτήν την οριμότητα της ε, ισπανικής κοινωνίας να αποτίσουμε φόρο τιμής. Για την δημοσιονομική εξηγένση μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία το 2011 η Ισπανική κυβέρνηση αντελήφθη, έμαθε, ότι είχε έλλειμμα 9,3% επί του ΑΕΠ η Ισπανική οικονομία. Καταφέραμε να το μειώσουμε στο 6,8% χωρίς ε, ε, την προσπάθεια αυτή, η διατήρηση των επιδομάτων ανεργίας που σημαίναν 5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, δαπάνη και ταυτόχρονα καταβολή των ε, επιπλέον ε, επιβαρύνσεων στον προπολογισμό στα 5 παλιδείς, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τις δαπάνες μας κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια με αύξηση φόρων που αποφασίστηκαν σε ύψος 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Τούτου λεχθέντος η προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση ήταν μια κίνηση απαραίτητη μια δράση απαραίτητη, γιατί είχαμε συστημικές δυσκολίες να χρηματοδοτήσουμε τον, τον κρατικό προϋπολογισμό και προκειμένου να περιορίσουμε τις οικονομικές πιέσεις χρειάστηκε να βοηθήσει και η ισπανική οικογένεια και σε αυτό θα πρέπει να απευθύνουμε τα εξή μήνυματα. Πρώτα απ' όλα ότι πρέπει κανείς να τακτοποιεί τα, τα, τα, οικονομικά του, όχι μόνο στην κεντρική κυβέρνηση αλλά και στις δαπάνες των περιφερειών και των τοπικών κυβερνήσεων και δεύτερον ή σε δεύτερο στάδιο να ε, προχωρήσουμε στις διαφορετικέ εκείνες μεταρρυθμίσει που θα εξασφαλίζουν μια υγιή οικονομία για το μέλλον. Πρόκειται δηλαδή για δύο, δύο βήματα παράλληλα και εξυγίανση και ταυτόχρονα υποστήριξη της μεσοπρόθεσμης, δυνατής μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαλντίνη, μέρος Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, θα είχα να θέσω πολλές ερωτήσεις, αλλά ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και η κυρία Μίλετιτς κάλυψε κάποιες από τις ερωτήσεις τις οποίες θα ήθελα και εγώ να θέσω. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, να συγχαρώ και την Ισπανία, γιατί έχετε προχωρήσει σε σημαντικές ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Σταθήκατε ικανοί να ανατρέψετε κάποιες αρνητικές τάσεις στην ισπανική οικονομία και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα εδώ σχετικό με κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες χώρες και για την νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δική μου χώρα την Κροατία. Ε, και η περιοχή αυτή διέρχεται μια δύσκολη οικονομική κρίση. Και είχα τρεις ερωτήσεις αρχικά, αλλά τις έχετε καλύψει και θα περιοριστώ μία. Θα ήθελα να μάθω αν η Ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει την διακυβερνητική αντιμετώπιση του προβλήματος σχετικά με το Ταμείο Εξυγίανσης. Και σε αυτή την περίπτωση γιατί πιστεύετε ότι η επιλογή αυτή από ότι εάν είχε ακολουθηθεί η κοινοτική μέθοδος. Well, respect to σχετικά με την διακυβερνητική διάσταση στην οποία αναφερθήκατε, θα πρέπει να πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει αυτή την διακυβερνητική πρόταση για, για αλλαγή της συνθήκης. Για ποιο λόγο τώρα. Γιατί πιστεύουμε ε, ότι από τις υπάρχουσες λύσεις ήταν η καλύτερη, δεν είναι η ιδανική αλλά ίσως είναι η μόνη η οποία είναι πραγματικά διαθέσιμη έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα των, των, τραπεζών. Όπως έχω ήδη πει, καταλήξαμε σε μια ευαίσθητη αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματική συμφωνία στο Συμβούλιο για τις Τράπεζες. Όλοι έπρεπε να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, και νομίζω ότι το χειρότερο σενάριο για όλους θα ήταν να μην υπάρξει μια τέτοια συμφωνία για την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων των τραπεζών. Και κάτι το οποίο θα υπονόμευε το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωζώνης. Γι' αυτό ακριβώς θελήσαμε να είμαστε επικοδομητικοί έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία. Είδαμε και το τι εναλλακτικέ λύσεις ε, υπήρχαν. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος να αντιμετωπίσουμε την συμφωνία αυτή με διακυβερνητικό τρόπο. Ο κύριος Λούις Δεγκράντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να πω ότι είσαστε μεν μετριοπαθείς, αλλά θα είχατε δίκιο να είσαστε και υπερήφανος, γιατί ε, αυτός ο οποίος αλλάζει ε, την βαθύτατα την ε, ισπανική οικονομία, ταυτόχρονα παρουσιαστήκατε εδώ επανειλημμένα, αυτοί οι οποίοι δημιουργούν σήμερα, λειτουργούν αρνητικά, είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν την Ισπανία στο παρελθόν στην δύσκολη φάση την οποία αντιμετώπισε. Νομίζω ότι ο δρόμος τον οποίο επιλέξαμε είναι πάρα πολύ δύσκολος αλλά απαραίτητος. και σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι φωνές να λέγουν ακριβώς από την υπόλοιπη Ευρώπη στα ε, θετικά για τα αποτελέσματα στα οποία εσείς είσαστε πρωταγωνιστής αλλά φυσικά πρωταγωνιστής ήταν και η κοινωνία της ε, Ισπανίας η οποία έκανε τεράστιες ε, θυσίες βέβαια αλλά και εσείς κάνατε κάθε προσπάθεια. Ο κύριος Μπαρότο έλεγε σωστά ότι η πολιτική διαλεκτική έριχνε θεωρητικά το βάρος στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αρνητικά και όλα τα θετικά στους υπόλοιπους. Νομίζω λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε creo que Νομίζω ότι είναι κουραστικό να ακούει κανείς την ισπανική αντιπολίτευση η οποία έχει μία φωνή μετριοπαθή αλλά και άλλες εκφράσεις ιδιαίτερα ακραίες να εξηγούν πάρα, με υπεραπλουστευμένο τρόπο την σημερινή κατάσταση και δείχνει ακριβώς την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η Ισπανία σήμερα είναι ένα σωστό παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία χώρα μέλος. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήσιμη, είναι ικανή να βοηθήσει σε περιπτώσεις ε, δύσκολες και επικίνδυνες μέσω ακριβώς αυτής της συμβιωτικής αντίληψης. Σας εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο. θα ήταν ε, πραγματικά συγχώρητο το να μην προχωρήσει κανείς σε αυτά τα δύσκολα θέματα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και μικροοικονομικά θέματα. Κατανοώ ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ο πρόεδρος Σούλτς, ο οποίος είναι υποψήφιος, είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των τραπεζών και με διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω τι είδους παρατηρήσεις, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τις παρατηρήσεις. Αλλά μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική σπάνια για την Ισπανία το θέμα είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε τα θέματα της μακροοικονομίας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν, ε, θα, δεν μειώνει τις θυσίες της κοινωνίας και γι' αυτό τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ε, της, ε, στον τομέα της απασχόλησης, τι μέτρα εν πάση περιπτώσει θα πάρει για να ευκολύνει εν πάση περιπτώσει να διευκολύνει τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες απαιτούν θα έλεγα δράση από πλευράς της ισπανικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για την φορολογική μεταρρύθμιση, τη μεσογειακή μεταρρύθμιση στην εγκρίνη κυβέρνηση που θέλουμε να δώσουμε όθηση με αυτήν ε, στην αποταμίευση, επενδύσεις, μικροσφαίρες επιχειρήσεις, από απασχολούμενους, να άρουμε πολλά από τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να ε, απλουστεύσουμε, να διευκολύνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. την είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Δεύτερον, βέβαια, πρέπει να εγκρίνουμε την ε, σχετική νομοθεσία για τα επαγγέλματα και κυρίως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν ε, το διοικητικό κόστος ε, και τα άλλα διοικητικά εμπόδια ώστε να μπορέσουν επαγγελματίε ε, να ωφελήσουν και τους τελευταίους, τους δελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών τους που είναι οι καταναλωτές, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης η κυβέρνηση θα εγκρίνει τις επόμενες ημέρες ε, έναν ε, χρηματοοικονομικό νόμο που θα έχει να κάνει με το κεφάλαιο πιωματικού κινδύνου για να έχουμε όλο και πιο πολλές επενδύσεις κεφαλαίου για επανακεφαλαιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διάφορα, άτομα, ε, διάφορα ταμεία όπως το Φόντο Διενβερσίων φακτούρας είχαμε καθυστέρηση πληρωμών σε διάφορους τομείς και αυτό είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Επίσης, προωθούμε και εναλλακτικούς τρόπους τραπεζικής χρηματοδότησης, όπως είναι οι υποσχετικές και τα λοιπά. Τέλος τους τελευταίους τρεις με έξι μήνες θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας ε, στον τομέα της φορολογίας. Είναι νομίζω ε, σαφές από όλους μας ότι έχουμε πρόβλημα ίσπραξης φορολογικών εισόδων και σίγουρα μπορεί το φορολογικό σύστημα να βοηθήσει να ανακάμψει η οικονομία, να έχουμε απελευθέρωση, να έχουμε εξάλληψη των ε, εμποδίων. Πρόεδρος εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για μια ακόμη φορά ο κύριος Σάντσεθ Πρεσέδο. Αφήστε όμως και ένα λεπτό να απαντήσει ο Υπουργός αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή οικονομία, ότι είναι ανεμική, είναι εύθραυστη, ε, λέγονται αυτά, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε προς μια ευρωστή οικονομία, ισχυρή οικονομία. Και να μην ε, βάλουμε σε κίνδυνο μια γενιά ολόκληρη από νέου. Δεν θέλω να κάνουμε εσωτερική συζήτηση νοισπανική, αλλά πώ μπορεί η να βελτιώσει την γενικότερη ευρωπαϊκή απάντηση. Λοιπόν, έρχομαι στα εξαιρετικά Πρώτον, ε, Τραπεζική Ένωση λέει το δούνο του ότι χρειάζεται από την πρώτη στιγμή να είναι επιχειρησιακή αυτή η Τραπεζική Ένωση. αυτό το ταμείο, ε, γιατί το Συμβούλιο δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, δηλαδή το δεσμευμένο κεφάλαιο φενό ε, και το εκταμιευθέν από την άλλη. Δεύτερον, ε, ω συνομοθέτε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να προωθήσει μια συμφωνία και τρι... διακυβερνητική συμφωνία και τρίτον. Πρέπει να έχουμε αξιοπιστή και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Και τι γίνεται με αυτό το δίκτυο ασφαλείας Τώρα, βελτίωση των ισολογισμών. Το δουν του λέει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων, των μη χρηματοπιστών επιχειρήσεων, για να δοθεί νέα όθηση στην ανάπτυξη. Πώ μπορεί να γίνει αυτό όμω, και πού μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, βιωσιμότητα του δημόσιου χρέου. Πρέπει να φέρει σε πέρα πολιτικές της η Ισπανία και στην Ευρώπη πρέπει να, γίνουν, να υπάρξουν αναπτυξιακά μέτρα πρέπει να υπάρχει ταμείο εξαγοράς του χρέους για το δημόσιο χρέος, ώστε να είναι βιώσιμο. Τέταρτον, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν βέβαια επενδύσεις. Ε, άρα πρέπει να έχουμε πρότυπα, κανόνες για την εκταμείωση πόρων προς τα κράτη-μέλη. Πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της σύγκλησης και της ανταγωνιστικότητας. Απαιτούνται νέα εργαλεία στην Ευρωζώνη και στην ε, ΟΝΕ. Και άλλη πτυχή σημαντική φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι άκρος σημαντικό. Μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα την οικονομική και στον ισομερή επιμερισμό των βαρών. Γιατί να πληρώσουν το τίμημα οι καταναλωτές. Αυτά θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σχετικά με την Τραπεζική Ένωση. Οι χώρες είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν πρώτα τα προβλήματα των τραπεζών. Το σύστημα, αν θέλετε, ε, λειτουργεί μέσω της ορολογίας που χρησιμοποιούμε του bail-in, αν μια τράπεζα έτσι και αλλιώς χρειάζεται κεφάλαιο, περνάει από διαφορετικά στάδια για να το αποκτήσει και από κάποια στιγμή και μετά τίθεται σε λειτουργία ο κοινό μηχανισμός ε, αντιμετώπισης των προβλημάτων των ε, τραπεζών. Η, Ισπανία θα είναι ίσως η τρίτη χώρα που θα συνεισφέρει, ίσως θα καλύψουμε το 16%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 θα δοθούν χρήματα λοιπόν στις τράπεζες, θα δίδονται χρήματα στις τράπεζες οι οποίες θα έχουν ε, ζητήσει και θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μοναδικό μέσο το οποίο βέβαια θα έχουμε στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε γρήγορα ε, στα θέματα των πιστοτικών προβλημάτων. Κάποιες εναλλακτικές λύσεις είχαν ίσως ακουστεί, αλλά Σίγουρα το σύστημα αυτό, ναι μεν δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο θα λύσει τα προβλήματα με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Υπακούει η, η βιωσιμότητα αυτή σε διάφορους παράγοντες. Εξαρτάται από το ονομαστικό επίπεδο, εξαρτάται από το ύψος των επιτοκίων Μείωσε το κόστος Μειώθηκε το μέσο κόστος έκδοση ομολόγων, ε, τα επιτόκια δηλαδή. Δεύτερον, μείωση δημόσιου χρέους για να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι κάτι που νομίζω μπορούμε να το πετύχουμε το 2016 και είναι θετικό για να μελλοντικό μονοπάτι θα ακολουθήσουμε για το δημόσιο χρέος και τέλο θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά ποσοστά ΑΕΠ. Στην Ισπανία, στην κρίση, ε, το output έπεσε 7 μονάδες ε, και γι' αυτό και το ονομαστικό ΑΕΠ ε, έπεσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δείτε αυτή την αναλογία και με τη βιωσιμότητα, δεν είναι μόνο, επειδή έχουμε, μιλάμε για ένα λόγο και ο, αριθμητής και ο παρονομαστής πρέπει να εξελίσσονται να βελτιώνονται για να πετύχουμε τη βιωσιμότητα. σε μεταρρυθμίσεις συμφωνώ μαζί σας με τα κοινοτικά εργαλεία που είπατε, αυτό το σχέδιο για την ενική απασχόληση και στο ΕΚΟΦΗΝ το είπαμε ότι έχουμε ένα δις και με τις αυτόνε περιφέρειες θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια και των διαθετικών ταμείων η έρευνα και ανάπτυξη, σημαντικό θέμα. Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, Ισπανία, συμμετέχει σε ενισχυμένη συνεργασία με άλλες χώρες, δέκα ακόμη χώρε και αυτό πρέπει να ορίσουμε και είμαστε σε αυτή τη φάση και ελπίζω του επόμενους μήνες να έχουμε σαφή αποτελέσματα είναι το εύρος του φόρου αυτού. Θέλουμε να παράγει μεν πόρους, αλλά να μην δημιουργεί και στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τα χρηματοψηφιακά ταμεία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. τελευταίο ο κύριο Τόρβαλ, μέσα των φιλελευθέρων. Και βέβαια θα μιλήσω και εγώ μετά τελευταίο ο εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Λυπούμε που καθυστέρησα και δεν μπορούσα να σα ακούσω από την αρχή. Είχαμε ένα θέμα με το Ταμείο αλία και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον μακροπρόθεσμα την ε, Ισπανική αλία. Ακούσατε όλα τα συγχαρητήρια, δεν θα τα επαναλάβω. Βλέπουμε κάποια εσπεράντσα, όπως τα λέγατε και εσείς Ισπανοί, κάποια ελπίδα στον ορίζοντα. Τις τελευταίες εβδομάδες ταξιδεύουμε, επισκεπτόμαστε τις ε, χώρες ε, των οικονομικών προγραμμάτων, των μνημονίων. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση αυτό που διαπιστώνουμε λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικά ευρωπαϊκά μέτρα για τη βελτίωση τη ευρωπαϊκής αλυσίδας αξιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και στην Πορτογαλία όπως και στην Ελλάδα και σε ένα βαθμό και στην Ισπανία. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική. Επίσης, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική ανάπτυξη είναι αλληλένδετα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια και στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα των γυναικών. Θεωρείτε ότι έχετε βρει τη σωστή λύση για τα δικαιώματα των γυναικών σε συνδέσμο με την οικονομική ανάπτυξη και αυτό γιατί καταλαβαίνετε ασφαλώς ποιο είναι το πνεύμα της ερώτησής μου. Να κάνω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις ε, γιατί πράγματι είχαμε προβλήματα με την ανταγωνιστικότητα και αν η βελτίωση του ισοζύγου πληρωμών είναι κάτι δομικό ή συγκυριακό. Έχετε το λόγο. Πολύ γρήγορα, σε σχέση με την ερώτηση σας. Σε ένα σημείο ίσως ε, θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε ότι παραβλέψαμε ένα θέμα στο προγράμματα διάσωσης. Αυτό το λεγόμενο ownership, την αποδοχή δηλαδή από τους πολίτες των μέτρων και των προγραμμάτων αυτό το αίσθημα αποδοχής μέτρων σκληρών που χρειάστηκε να πάρουν ε, κάποιες χώρες ή που επιβλήθηκαν έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία. Εδώ το... Ε, η, η εξίσωση έχει αρνητικό πρόσημο και πρέπει στο μέλλον να το αποφύγουμε αυτό το έλλειμμα. Για τη δεύτερη σας ερώτηση η Ισπανία πιστεύω θα προχωρήσει και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην οικονομία. Είναι σημαντικό βεβαίω να έχουμε οικονομική πρόοδο. Αλλά και οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα όντα έχουν μεγάλη σημασία και σε αυτά θα πρέπει να εστιαστούμε. Στην ευημερία των ανθρωπίνων όντων σχετικά με τα θέματα της ανταγωνιστικότητας. Είναι ένα θέμα αρκετά νέο και δύσκολο. Το τι στάση θα κρατήσουμε στο προσεχές μέλλον και τι αναλύσεις μπορούμε να κάνουμε στην ζώνη ερώ. Το θέμα είναι πώς μπορεί να εκφραστεί η ανταγωνιστικότητα σε μια νομισματική ένωση. Ε, υπήρχαν στο παρελθόν δυνατότητες να ελεγχθεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας και με τις νομισματικές πολιτικές, με τις ισοτιμίες, με τις πραγματικές ισοτιμίες, με τις αυξήσεις των ε, εξαγωγών, αλλά υπήρχαν βέβαια και πλάγιες παράπλευρες επιπτώσεις όπως ο πληθωρισμός. Αυτό επηρέαζε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Στην Ισπανία τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, καταρχάς το εργασιακό κόστος, του ελέγχου του μισθολογικού κόστους, βλέπουμε εμείς να έχουμε χαρακτηριστικά θετικά στον τομέα της παραγωγικότητας μέσω μιας καλύτερης ευελιξίας της αγοράς εργασίας και μέσω της γενικότερα καλύτερης ανταγωνιστικότητας της ισπανικής οικονομίας και ευελιξίας. Αυτό σημαίνει και έλεγχος του πληθωρισμού. Εδώ ο πληθωρισμός είναι 0,3%. και αυτό αφορά και τον συνολικό ε, πληθωρισμό που μπορεί να φτάσει συνολικά το 0,5. Αυτό είναι θετικά και για τους καταναλωτές και θετικό συνολικά για την επόμενη φάση γιατί μπορεί έτσι να υπάρξει δυνατότητα αύξησης των οικονομικών δυνατοτήτων των εργαζομένων. Εμείς είδαμε στα πλαίσια των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όλοι οι αναλυτές ε, ακούγεται ότι οι προβλέψεις του για τα επόμενα 3-4 χρόνια λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Αλλά πάντως είναι σαφές ότι η Ισπανία θα έχει πλεόνασμα τα επόμενα έτη και αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό της εξυγίανσης της ε, ισπανικής οικονομίας. Αυτή η φούσκα στο πιστοτικό σύστημα που είχαμε στο παρελθόν θα απαλλαγούμε από αυτή. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα λοιπόν επιβίωσης της ε, ισπανικής οικονομίας δείχνει ότι ε, θα υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης έτσι ώστε η Ισπανία εκ νέου να βρεθεί σε μια θέση η οποία να επιτρέψει την οικονομία της να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό Είναι μία από τις τελευταίες ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια αυτής της εντολής που τον συναντάμε και θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει. Disculpen, la próxima reunión será el jueves a las 9 eh, de la mañana hasta las 12 y media. Gracias. Πέμπτη στις 2.30 λοιπόν, από τις 9 το πρωί και μετά στις 2.30.